Λοιπόν, θα συνεχίσουμε ε, με τις επεξηγήσεις ψήφου τώρα. Θα παρακαλούσα όλους όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το πράξουν ησύχως. Καλό σας ταξίδι, καλή σας όρεξη αναλόγως. Ευχαριστώ πολύ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 Το πρώτο θέμα είναι οι τρίτες χώρες υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Είναι η έκθεση Αγκουστίν Δίας Δεμέρα Γκαρσία Κοσουέγρα. Η κυρία Μακοβέη, κυρια μακοβεη θέλω για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο μηχανισμός αυτός ε, αναστολής της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίων ε, για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστεί πολύ